Allora, Ο έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ για την ε, καλοσύνη σας και για την πρόσκλησή σας. Ε, θα συνεχίσω στα αγγλικά με την άδειά σας. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία αυτή να σας παρουσιάσω το όραμά μου και τις ε, φιλοδοξίες μου για τη θέση του ε, Ευρωπαίου Διάσημου Μεσολαβητή. Έχω υποβάλει σε 23 γλώσσες ε, το βιογραφικό μου σημείωμα, το οποίο τονίζει τα βασικά προσόντα που φέρνω στη θέση αυτή. Καταρχήν η επαγγελματική μου εμπειρία ως συνήγορος του πολίτη στην Ελλάδα και ως Ευρωπαίο Μεσολαβητή μετά τον Απρίλιο του 2003 Τέλο ε, την ε, ανεξαρτησία μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα 225 μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τα 27 κράτη-μέλη που ε, επιβεβαίωσαν την υποψηφιότητά μου για να ξαναυποβάλω υποψηφιότητα. Αποτελεί τιμή για μένα το γεγονό ότι τόσοι βουλευτέ από τόσε διαφορετικέ πολιτικέ ομάδε με υποστήριξαν μια τέτοια ευρεία υποστήριξη αποτελεί ε, μια σημαντική ε, υποστήριξη για τον ε, Ευρωπα... νομιμοποίηση για τον Ευρωπαίο διαμεσολαβητή στα μάτια του Ευρωπαίου πολίτη. Διαμεσολαβητή θα ήθελα του Ευρωπαίου πολίτη, συγγνώμη. Θα ήθελα να σας αναφέρω τα επιτεύγματά μου. Καταρχήν, μια πιο αποτελεσματική προσφυγή για τους πολίτες σε περίπτωση που δεν ε, ε, γίνονται σεβαστά τα δικαιώματά τους και η μεγαλύτερη διαφάνεια. Με τις ε, έρευνες πρωτοβουλία μας αλλά και με τις απαντήσεις στις προσφυγές έχω βελτιώσει τις βέλτισες πρακτικές με τις ετήσιες εκθέσεις μου όπου δίνω παραδείγματα της καλής διακυβέρνησης Έχουμε λύσει ε, προβλήματα ε, καθυστερημένων πληρωμών, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους ε, μεμονωμένους πολίτες. Επίσης, έχουμε ασχοληθεί με την υπερβολική γραφειοκρατία, ιδιαίτερα εις βάρος των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Έχουμε βελτιώσει την διαδικασία επιλογής της ΕΠΣΟ, και ως αποτέλεσμα το 2008 40% λιγότερες προσφυγές κατά της ΕΠΣΟ είχαμε από ότι το 2007. Έπεισα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανταποκρίνονται σε αιτήματα των πολιτών και να λαμβάνουν υπόψη την προοπτική του πολίτη όταν λαμβάνουν αποφάσεις. Επίσης έκανα αυτά που έλεγα. Ε, προσπάθησα να ε, θέσω ένα καλό παράδειγμα όσον αφορά την υπηρεσία προς τον πολίτη, ιδιαίτερα η υιοθέτηση. Υιοθέτησα νέο σαφή μορφότυπο για τις αποφάσεις και ε, επίσης εκπαιδεύσαμε στα απλά αγγλικά το προσωπικό μας για να είναι πιο κατανοητές οι αποφάσεις. Πάνω από 200 ομιλίες έκανα για να γνωρίζουν οι πολίτες τα δικαιώματά τους ε, όσον αφορά τις προσφυγές. Επίσης, είχαμε καλή ε, διακυβέρνηση όσον αφορά τον προϋπολογισμό στην οργάνωση του φορέα μας. Ε, αναδιοργανώσαμε την ιστοθέση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για να είναι ελκυστική και κατανοητή σε 23 γλώσσες. Την ετήσια έκθεση την κάναμε πιο σύντομη, πιο επικεντρωμένη στα βασικά θέματα και πιο φιλική προς αναγνώστη. Επίσης, ε, βελτίωσα την ε, πρόσβαση στις πρόσφυγες για τους πολίτες ε, και σε επίπεδο ένωσης χρησιμοποίησαμε πιο γρήγορες και ευέλικτες διαδικασίες. Έχουμε συντομεύσει το χρόνο για τη λύση των προσφυγών και έχουμε εκδώσει έναν οδηγό που βοηθάει τους ε, πολίτες, στις ε, επιχειρήσεις και τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Ο οδηγός αυτός ήδη έχει χρησιμοποιηθεί από πάνω από 24.000 πολίτες από ε, την έκδοσή του φέτος τον Ιανουάριο. Με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων υπογράψαμε μνημόνιο κατανόησης. Η τράπεζα έχει βελτιώσει το σύστημα προσφυγών της Επίσης, ε, ξεκινήσαμε ετήσιες ε, μελέτες ε, και χρησιμοποίησα τις ενισχυμένες αρμοδιότητες που μου έδωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε επίπεδο κρατών μελών συνεργάστηκα με εθνικούς και περιφερειακούς διαμεσολαβητές για να ενισχύσω το ευρωπαϊκό δίκτυο διαμεσολαβητών για να εξυπηρετήσουμε τους πολίτες στις διάφορες περιφέρειες. Η συνεργασία αυτή βελτιώθηκε με πάνω από 100 επισκέψεις σε όλα τα κράτη-μέλη, όπου συνάντησα πολίτες, δημόσιες διοικήσεις, την κοινωνία των πολιτών, μέλη των κυβερνήσεων και το δικαστικό σώμα. προώθησα την υιοθέτηση μιας δήλωση από όλα τα μέλη του δικτύου όσον αφορά την, τις υπηρεσίες που προσφέρουν στους πολίτες. Βελτίωσα τις ε, υπηρεσίες συμβουλών προς τους εθνικούς συνηγόρους του πολίτη που έχουν απορίες σχετικά με το ε, δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ερμηνεία τους. Έτσι βοηθάμε τα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν σωστά το ε, δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, ενθαρρύναμε την καλή επικοινωνία ανάμεσα στους διαφόρους συνηγόρους του πολίτη και το δίκτυο Solvit. Σύμφωνα με τον κανονισμό 1041 του 2001, προωθήσαμε την ε, διαφάνεια, βελτιώσαμε την πρόσβαση των πολιτών στα ε, έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατόπιν ε, συμφωνία και μάλλον υπογράψαμε μνημόνιο κατανόησης με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή για την προστασία των δεδομένων. Αναπτύξαμε επαφές με εθνικούς ε, επιτρόπους για την πληροφόρηση στα κράτη-μέλη, ε, ε, θέτοντας έτσι τις βάσεις για τη μελλοντική συνεργασία. Γενικά κατάφερα να βοηθήσω το 80% των ανθρώπων που προσέφηκαν σε μένα είτε άμεσα είτε παρέχοντάς τους πληροφορίες σχετικά με το που μπορούν να στραφούν σε περίπτωση που δεν μπορούσα να ξεκινήσω εγώ έρευνα. Οι δραστηριότητες πρωτοβουλίας μου ε, ε, ε, βοήθησαν στο διπλασιασμό της κάλυψης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Διαμεσολαβητή και στην υποβολή σημαντικών υποθέσεων για θέματα αρχής, θέματα που είχαν να κάνουν με τα δικαιώματα υπεράσπισης, την κατάχρηση εξουσίας κλπ. Σύμφωνα με το Ευρωμάτρο του Μαΐου 2008, το 38% των Ευρωπαϊκών πολιτών γνωρίζουν τι είναι ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής. Έχουν ακουστά το Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Αυτό είναι πολύ ικανοποιητικό νούμερο, δεδομένου ότι η εντολή του διαμεσολαβητή περιορίζεται στα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τις υπηρεσίες τους. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα ήταν δυνατό χωρί ε, την συνεργασία του ε, Κοινοβουλίου το Κοινοβούλιο μου έδωσε το δυναμικό που χρειαζόμουν για να κάνω τη δουλειά μου και η Επιτροπή σας ασχολήθηκε ε, αποτελεσματικά με θέματα στα οποία επέστρεψα την προσοχή σας. Ιδιαίτερα όσον αφορά τις ειδικέ εκθέσεις που θεώρησα ότι είναι απαραίτητο να υποβάλω. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές. Σίγουρα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συχνά θεωρούνται απόμακρα και απρόσωπα μία απρόσωπη γραφειοκρατία. Ωστόσο, είμαι βέβαιος ότι υπάρχει ε, συμφωνία μεταξύ μας ότι η διατήρηση υψηλής ποιότητας ε, στην ε, διοικητική πρακτική όχι μόνο θα ωφελήσει τους πολίτες, αλλά θα λύσει σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα αυτά. Είμαι περήφανος για τα αποτέλεσματα που έχω πετύχει ως διαμεσολαβητής, ωστόσο γνωρίζω ότι Υπάρχουν πολλά που πρέπει και μπορούν να γίνουν ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν απόλυτα τα δικαιώματά τους ε, και πώς μπορούν να τα ασκήσουν. Είναι σαφές από τις απαντήσεις ε, των θεσμικών ε, οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις έρευνές μου ότι ήδη υπάρχει υψηλό επίπεδο διοικητικής πρακτικής. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι ο αριθμός των υποθέσεων για την ε, κακή διαχείριση είναι πολύ λίγε. Μόνο 16 ειδικέ εκθέσεις έπρεπε να υποβάλει ο διαμεσολαβητής σε 14 χρόνια λειτουργία του. Ωστόσο, οι βελτιώσεις μπορούν και πρέπει να γίνουν από τις υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να ε, δημιουργηθεί μια κουλτούρα υπηρεσίας προς τον πολίτη. Ένα τέτοιο στόχο μπορεί να βοηθηθεί από έναν διαμεσολαβητή που είναι απόλυτα ανεξάρτητο και δίκαιο και αμερόληπτος. Αυτός είναι ένας στόχος τον οποίο έχω επιδιώξει συστηματικά στα χρόνια που, της θητείας μου και που θα συνεχίσω να επιδιώκω εάν επανεκλεγώ. Όπως ε, ήδη ε, έχω πει στις ε, απαντήσεις μου σε ερωτήσεις που στείλατε σε όλους τους υποψηφίους και όπως ήδη έχει, αναγράφεται στην ιστοθέση του διαμεσολαβητή, ε, υπάρχουν τρεις προτεραιότητες ε, να διασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ωφελήσει τον πολίτη σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Δεύτερον, θα πρέπει να ενισχυθεί η κουλτούρα υπηρεσία στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέλος θα πρέπει να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της θέσης του ε, Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Επιτρέψτε μου να αναπτύξω τις ιδέες που ανέφερα στις γραπτές μου απαντήσεις κύριο στόχο των ε, θεσμικών οργάνων τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι να ε, καταστήσουν επιτυχία την ε, συνθήκη τη Λισαβόνα και να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του πολίτη. Η συμβολή του διαμεσολαβητή θα πρέπει να είναι ότι οι πολίτε θα αποφελούνται από την καλή διοίκηση και ότι θα γνωρίζουν τι διατάξει τη συνθήκη όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματά του και να έχουν πρόσβαση σε έγγραφα, να μπορούν να προσφύγουν στον ή στο κοινοβούλιο ώστε να μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους. Στοχεύω να επικαιροποιήσω τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Καλής ε, Διοικητικής ε, Πρακτικής ε, υπό το φως των βέλτιστων πρακτικών που έχει αναπτύξει ο διαμεσολαβητής και άλλοι και την ε, διοικητική νομολογία και την ε, συνθήκη της Λισαβόνας, ώστε τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υιοθετήσουν τον κώδικα αυτό και να τον ακολουθούν όσο γίνεται. Θέλουμε να αναπτύξουμε την ε, δυνατότητα ερευνών πρωτοβουλίας. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα άτυπο δίκτυο καλής διοίκησης, να μοιραζόμαστε τις βέλτιστες πρακτικές, να παρέχουμε κατάρτιση, να συνεργαζόμαστε στενά με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους φορείς τη, ώστε να διασφαλίσουμε τις φιλικές λύσεις. Θέλουμε να συνεργαστούμε στενά με την Επιτροπή αυτή και με το Κοινοβούλιο στο σύνολό του. Επιπλέον, προτείνω στο νομοθετικό διάλογο να έχω μια πιο ε, ισχυρή θέση, να παρεμβαίνω στις δημόσιες συζητήσεις όσον αφορά την προτινόμενη νομοθεσία για θέματα που αφορούν τον ε, διαμεσολαβητή, όπως είναι ε, ο κανονισμός για τον Όλαφ, ο δημοσιονομικός κανονισμός κλπ. Εάν με επανεκλέξετε, προτείνω να κάνω τα εξής. Να ενισχύσω τις επαφές με εθνικούς φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ώστε να διασφαλίσουμε τις βέλτιστες πρακτικές και την, την καλύτερη πληροφόρηση. Να συνεργαστώ με τα κράτη-μέλη για την οργάνωση εκδηλώσεων που θα χρησιμοποιούν την εμπειρία του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Επίσης ε, θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε του φορεί πληροφόρηση του Κοινοβουλίου για να ενημερώσουμε καλύτερα του πολίτε. Τακτικά να οργανώνουμε εκδηλώσεις ε, μαζί με, σε συνεργασία με ενδιαφερομένους ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να δημιουργήσουμε ένα, φόρουμ, ένα συνεχές φόρουμ για διάλογο με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την κοινωνία των πολιτών. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ε, ιστοθέσεις ε, κοινωνικής δικτύωσης ε, για να ερχόμαστε σε καλύτερη επαφή με τους πολίτες. Και τέλος θέλουμε να βελτιώσουμε την γνωστική βάση των του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών και Παρομοίων Φορέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, η βελτίωση της ποιότητας ε, της διοίκησης προς όφελος του Ευρωπαίου πολίτη πάντα ήταν βασικός μου στόχος. Εάν με επανεκλέξετε θα υιοθετήσω ένα στρατηγικό σχέδιο για τη θέση του διαμεσολαβητή που θα έχει ως light motif ε, την εξής δήλωση. Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής επιδιώκει τις δίκαιες λύσεις σε προσφυγές κατά των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενθαρρύνει την ε, διαφάνεια και προωθεί μια ε, διοικητική κουλτούρα της υπηρεσίας. Θέλει να βελτιώσει την ε, εμπιστοσύνη μέσα από τον διάλογο με τους, Ευρωπαϊκ... τους πολίτες και την... τον διάλογο μεταξύ πολιτών και Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ε, οδηγηθούμε σε καλύτερα πρότυπα στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, θέλουμε μια διοίκηση με ανθρώπινο πρόσωπο που να είναι αφοσιωμένη στην ε, εξυπηρέτηση των πολιτών. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Θα ακούσω τις ερωτήσεις σας. Τώρα ανοίγει η συζήτηση. Γκρουνή, πρώτη παρέμβαση. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας κύριε Διαμαντούρο. Δεν θα επαναλάβω τις ερωτήσεις που σας υπέβαλα γραπτός, γιατί μας τις ε, ανακεφαλώσατε και στην απάντησή σας, στην εισήγησή σας μάλλον τώρα. Μέσα στα πλαίσια της θητείας σας θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο θα θέλατε να εφαρμόσετε κάτι που δεν μπορέσατε μέχρι τούδε. Έχετε νέους στόχους προσπραγμάτωση. Δεν φοβόσαστε να έχετε μία θητεία που θα είναι μία θητεία η οποία θα είναι μία παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε και πώς βλέπετε τη συνεργασία σας με τα άλλα θεσμικά όργανα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ευρωπαίοι Μεσολαβητή, είναι μεγάλη μου χαρά και ιδιαίτερο πλεονέκτημά μου να σας καλωσορίσω εδώ στην ακρόαση αυτή. Με στενή συνεργασία με την Επιτροπή μας του Ευρωπαϊκού Διαμεσολαβητή, οι πολίτες μπορούν πλέον να δουν καλύτερα ποια είναι η διαφορά μεταξύ καλής και κακής διαχείρισης και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάτι το οποίο θα πρέπει να προωθήσουμε περαιτέρω. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, είστε διατεθειμένος να συνεργαστείτε για ένα κοινό μηχανισμό αντιμετώπισης των αναφορών προκειμένου να βελτιωθούν οι σχέσεις μεταξύ Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ. Ε, Κύριε Διαμαντούρε, να σας ζητήσω συγγνώμη γιατί θα επαναληφθώ ως ένα βαθμό. αλλά στις γραπτές σας, στη γραπτή σας εισήγηση, αλλά και στα προφορικά σας σχόλια, περιλαμβάνεται ένα σημείο το οποίο με απασχολεί ιδιαίτερα. Δεν το βρήκα όμως στην παρουσίασή σας στο σημείο αυτό, το θέμα των δικαιωμάτων των εθνοτικών μειονοτήτων. Δεν ήμουν ίσως σαφής προηγουμένως, δεν έδωσα παραδείγματα, θα δώσω παραδείγματα. Μπορεί σε ένα κάποιο κράτος μέλος ο νόμος να προβλέπει ότι οι εθνικές ε, μειονότητες δεν μπορούν για παράδειγμα να χρησιμοποιήσουν την εθνική τους γλώσσα. Την γλώσσα τους. Μιλάμε για μια συλλογική παραβίαση δικαιωμάτων. Αλλά και παραβίαση των ατομικών δικαιωμάτων του κάθε ανθρώπου που προκαλεί προσωπικά πόνο σε κάθε άτομο. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε, τι μπορείτε να κάνετε εσείς, τι θεωρείτε ότι μπορεί να γίνει γενικότερα για να διορθωθεί η κατάσταση αυτή. Πώς μπορούμε να βρούμε μια έναν ειρηνικό τρόπο επίλυσης των διαφορών αυτών. Χωρίς να αγνοούμε τις παραβιάσεις αυτές, χωρίς να κάνουμε ότι δεν υπάρχουν, πρόκειται για παραβιάσεις που επηρεάζουν τόσο ολόκληρες ομάδες, αλλά και μεμονωμένα άτομα του πληθυσμού. Τα δικαιώματα των μειονοτήτων είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί, κάτι το οποίο όμως θα πρέπει να κοιτάξουμε και περισσότερο σε πιο αφρημένο επίπεδο, αν θέλετε. Το θέμα αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο γιατί θέλουμε να επιλύσουμε συγκεκριμένες διαφορές, αλλά και επειδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργείται μια αίσθηση αγανάκτησης, ότι κάποιους ανθρώπους τους παρατάμε δηλαδή. Και έχει ο κόσμος την αίσθηση ότι εφαρμόζουμε διπλά μέτρα και σταθμά. τα προβλήματα αυτά ανακύπτουν σε απομακρυσμένες γεωγραφικά περιοχές. Αυτό δεν αποτελεί από μόνο του πρόβλημα, αλλά δεν καταλαβαίνει ο κόσμος γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφεύγει να αντιμετωπίσει τέτοια προβλήματα. Αν και η παραβίαση των ατομικών αυτών δικαιωμάτων σημαίνει και η παραβίαση των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάμε για την αξιοπρέπεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, σας ρωτώ, θεωρείτε ότι υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστούν αυτές οι παραβιάσεις και πώς θα καταργήσουμε τα διπλά μέτρα και σταθμά τα οποία εφαρμόζονται και σε πιο γενικό επίπεδο. Εσείς, πώς μπορείτε ως διαμεσολαβητής να εξασφαλίσετε ότι θα ευθαμιγραμμιστούν οι εθνικές και οι ευρωπαϊκές αρμοδιότητες για να μην υπάρχουν κρίσεις δομής. Thank you very much. Ευχαριστώ, κύριε Διαμαντούρε, κυρία Γκέντς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίασή σας. Ήταν πολύ συνοπτική και μιλήσατε και για τα μελλοντικά σας σχέδια. Σας ευχαριστώ γιατί ήταν μια ερώτηση που ήθελα να σας θέσω. Ποιες αλλαγές δηλαδή οραματίζεστε μετά την συνθήκη της Λισαβόνας και την ε, εφαρμογή της. Απαντήσατε όμως το ερώτημα αυτό, δεν χρειάζεται να το ξαναθέσω. Μία άλλη ερώτηση όμως, την οποία έθεσα και στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου. Μειώσατε σημαντικά τη διάρκεια χρόνου που αφιερώνεται στην απάντηση ερωτημάτων των πολιτών. Είναι ευαίσθητο το θέμα αυτό, ξέρετε, γιατί αν ο κόσμος έχει κάποια ερώτηση, θέλει να απαντηθεί η ερώτηση αυτή. Πώς θα αντιμετωπίσετε λοιπόν αυτό το θέμα της διάρκειας απάντησης των ερωτήσεων αυτών, γιατί νομίζω ότι είναι ένα θέμα που ανακύπτει συχνά. κυρία... Thank you very much. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Διαμαντούρο για την πολύ θετική παρουσίασή σας σε δύο πράγματα θα ήθελα να σας ρωτήσω. Καταρχήν, όλοι αναγνωρίζουμε την αφοσίωσή σας ε, στην ε, κουλτούρα υπηρεσίας στα θεσμικά όργανα. Πολλοί όμως ανησυχούμε ακόμα ότι οι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται αντιμετώπιοι με μια πληθώρα μερών όπου μπορούν να στραφούν, μπορούν ε, να στείλουν αναφορά στο κοινοβούλιο, μπορούν να στραφούν σε εσά, ε, μπορούν να ψάξουν στο Σόρβιτ, μπορούν να ε, ε, έρθουν σε επαφή με την Κομισιόν. Όλα αυτά μπερδεύουν τους πολίτες. Θα πρέπει να ενημερώσουμε τους πολίτες για το, για το πού πρέπει να στραφούν. Έχει αναφερθεί η λύση της ενιαίας θηρίδας ή μιας κοινή πύλης. Τι πιστεύετε εσείς. Δεύτερον, η μιας κοινης πυλης τι πιστευετε εσεις δευτερον η λισαβονα θα σημαίνει ότι το Συμβούλιο θα είναι ένα πολύ πιο σταθερό θεσμικό όργανο, θα παίζει σημαντικό ρόλο. Δεν ήταν όμως υπόδειγμα διαφάνεια τα τελευταία χρόνια. Πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό και τι θα γίνει με τα κοινοβούλια των κρατών μελών που πλέον θα συμμετέχουν στην νομοθετική διαδικασία. Προβλέπετε η ειδική σχέση με τα εθνικά κοινοβούλια και πώς βλέπετε τον πιθανό τους ρόλο ως νέο θεσμικό όργανο. Ευχαριστώ κυρία Όκεν. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη δουλειά σας και την παρουσίασή σας. Νομίζω ότι πολλές από τις ερωτήσεις μας μοιάζουν με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Θα έχουμε δύο νέα άρθρα που προσφέρουν νομική βάση για βελτίωση της διακυβέρνησης στα θεσμικά όργανα. Μιλήσατε γι' αυτό. Θα ήθελα να ακούσω συγκεκριμένα τι θα κάνετε γι' αυτό. Θα έχουμε κανόνες που να επιβάλλουν την καλύτερη διακυβέρνηση και επίσης όσον αφορά την παρακολούθηση των διαφόρων φορέων και θεσμικών οργάνων. Πώς θα βελτιώσετε την παρακολούθηση του τι συμβαίνει. Διότι νομίζω ότι αυτό θέλουμε να κάνετε και αυτό είναι πολύ κοντά στους πολίτες, διότι πολύ συχνά έρχονται σε επαφή με τις υπηρεσίες. Ευχαριστώ κύριος Τσίτσεστερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε καθηγητά, θα ήθελα να σας συγχαρώ για το βιογραφικό σας και την ε, πολύ ε, ενδιαφέρουσα παρουσίασή σας. Φαίνεται ότι ε, θέλετε πολύ να συνεχίσετε τη δουλειά που έχετε κάνει. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, τι θεωρείτε την, ποια θεωρείτε την καλύτερη μεμονωμένη απόφασή σας κατά τη διάρκεια της θητείας σας και δεύτερον ποια μεμονωμένη δράση ή απόφαση ε, έχετε μετανιώσει και θα ήθελα να ξέρω γιατί και στις δύο περιπτώσεις. Ε, στην γραπτή σας απάντηση αναφερόσαστε στην ε, θεσμοποίηση της παρακολούθησης της συνέχειας που δίνεται από τον διαμεσολαβητή σε υποθέσεις. Δεν είμαι βέβαιος ότι λάβαμε απάντηση σε αυτό. Εάν απαντήσατε, έχασα, θα ήθελα να αναπτύξετε το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ε, είχαμε την ευκαιρία πρόσφατα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συζητώντα την έκθεση της κυρίας Παλιαδέλη που είναι στο Δήμα, είναι στο Προεδρείο, να, ε, να εκτιμήσουμε και να αξιολογήσουμε κατά τη γνώμη μου θετικά το έργο του κυρίου Διαμαντούρου. Τον ευχαριστώ για την παρουσία του και για το έργο του και αξιοποιώντα τη σημερινή παρουσία του εδώ θα ήθελα να του υποβάλω ορισμένα ερωτήματα. Το πρώτο, από την εμπειρία του, τι προβλήματα συνάντησε με τους εθνικούς και περιφερειακούς διαμεσολαβητές και πώς τα έλυσε. Πώς πρέπει να λύνονται τέτοια προβλήματα. Το δεύτερο, μιλάει στη γραπτή απάντηση για την ανάγκη να προαχθεί και να παγιωθεί μια νοοτροπία εξυπηρέτηση του πολίτη στην Ευρωπαϊκή Δημόσια Δίκηση. Ξέρω ότι είναι μια δύσκολη, ένας δύσκολος στόχος. Όταν μάλιστα αναφέρεσε σε όργανα πολυσχηδή, αδιαφανή και κατά βάση μη ερετά. Εδώ κύριε Διαμαντούρο τι θα κάνουμε. Και το τρίτο για να μπορεί να προασπίσει, να, να γνωρίζει και να προσπίσει τα δικαιώματά του ο πολίτης πρέπει να τα γνωρίζει. Αλλά κατά την εκτίμησή μου η συνθήκη της Λισαβόνα, αλλά και ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων δεν είναι ευρύτερα γνωστός. Επομένως εδώ ποια κατά τη γνώμη σας, ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν κατά τη γνώμη σας για να μπορεί να γνωρίζει καταρχήν ο πολίτης τα δικαιώματά του, για να τα προασπίσει και να παραπέμπει ή να αναφέρεται σε εσά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σαλαβράκο. Κύριε είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω και εγώ τον απολογισμό του έργο σα και την έκθεση τη κυρία Παλιάδέλη, και πραγματικά ήταν εξαιρετικό. Οφείλω να το ομολογήσω. Όμω από αύριο αρχίζει μια καινούργια εποχή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εφαρμόζεται η συνθήκη τη Λισαβόνα και τα ίδια προβλήματα τα οποία θα υπάρξουν και για το κοινοβούλιο αυτό της αποτελεσματικότητας και της ουσιαστικής δηλαδή παρεμβάσεώς του στα βήματα της κοινότητας παρουσιάζονται για όλους τους παρεπόμενους θεσμούς μεταξύ των οποίων είναι και ο θεσμός του Όμπουσμαν. Πρέπει να διατηρηθούν ορισμένες πιστεύω αποτελεσματικές ε, και να διασφαλιστούν ορισμένες αποτελεσματικές παρεμβάσεις που αφορούν τόσο εμάς όσο και το θεσμό, του Όμπουσμαν. Έχετε επισημάνει εσείς πως ο θεσμός του Ευρωπαίου Μεσολαβητή εν ώψη της συνθήκης της Λισαβόνας και της εφαρμογής της θα γίνει πιο αποτελεσματικός για να μιλάμε πλέον σε ρεαλιστικό επίπεδο και όχι σε ένα επίπεδο ευχών ή ένα επίπεδο υπερβολικής ευγενίας και μη ρεαλισμού. Σας ευχαριστώ. Κύριος Διαμαντούρος έχει το λόγο για να ανταπαντήσει και μετά θα αρχίσουμε τη διαδικασία Catch the Eye. Grazie di Madame ah, je vous remercie beaucoup. Κυρία Γκρουνή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλιά σας. Είναι πάντα δύσκολο να απαντήσει κανείς σε μια ερώτηση τύπου μήπως κάνετε υπερβολικά πολλά. Δεν θα ήμουν υποψήφιος αν ε, είχα την εντύπωση ότι η θητεία αυτή θα ήταν μία ε, θητεία υπερβολικά, υπερβολική, δηλαδή μετά από την εξαετή μου θητεία. Νομίζω ότι προσπαθούμε να οικοδομήσουμε κάτι ως ε, διαμεσολαβητής. Προσπαθώ να χτίσω μία σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες. Πρόκειται για μία ε, μακρά και επίπονη διαδικασία. Γι' αυτό θεωρώ ότι εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με μου κάνει την τιμή να με επανεκλέξει διαμεσολαβητή, δια θα εμβαθύνω αυτά που ήδη έχω κάνει. Εσείς με ρωτήσατε κατά πόσο θα προσέβλεπα σε κάτι άλλο. Θα είμαι πολύ ειλικρινής. Ε, στα πλαίσια αυτής της προσέγγισης των πολιτών και της πληροφόρησης έχουμε να κάνουμε με έναν ε, μεγαλεπίβολο στόχο ο οποίος απαιτεί πολλές προσπάθειες και εγώ είμαι έτοιμος να το προσπαθήσω, βάση περιπτώσει. Βεβαίως υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης ενός στόχου. Οι μεγάλοι άξονες δεν μπορούν να έχουν μεγάλη ευρύτητα, γιατί πάντα με απασχολούν θέματα κακοδιοίκησης, διαφάνειας, καταπολέμησης των κακοδιοίκησεων, έτσι ώστε να προσεγγίσω αυτό το ζήτημα όσο το δυνατόν πιο σωστά. Για να απαντήσω σε μια άλλη σας ερώτηση, θεωρώ ότι η συνεργασία που προώθησα με την Επιτροπή Αναφορών διαχρονικά ήταν πολύ επικερδής και σημαντική για όλους. Ήδη προανέφερα ότι η επικύρωση συνθήκης της Λισαβόνας και η θέση της ισχύ από αύριο το πρωί είναι ύψης της σημασίας για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Διανοίγονται πολλές δυνατότητες έτσι ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορέσει να χρησιμοποιήσει την δυνατότητα συνεργασίας με τα εθνικά κοινοβούλια. Και επειδή εγώ ήδη διαθέτω ένα δίκτυο συνεργασίας με συνηγόρους του πολίτη σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο μπορώ να συνεργαστώ για θέματα καλής ή κακής διοίκησης έτσι ώστε να δράτω με τις ευκαιρίες κάθε φορά που μου παρουσιάζεται για να προωθήσω κάτι περισσότερο. Αλλά θα με βοηθήσει πάντα η υποστήριξη Επιτροπής Αναφορών, υποστήριξη την οποία πάντα είχα μέχρι τούδε. Βεβαίως, το θέμα συνεργασίας με τους άλλους φορείς ή με τους άλλους γενικότερα Εάν πρόκειται για τους εθνικούς ε, διαμεσολαβητές και τους περιφερειακούς ε, συνηγόρους ε, του πολίτη, θα χρησιμοποιήσω τη συνθήκη της Λισαβόνας για να ενισχύσω το δίκτυο του, των διαμεσολαβητών των κρατών μελών για να προχωρήσω πιο μακριά από ό,τι καταφέραμε μέχρι του παρόντος. Αυτό το οποίο είναι φοβερό και ελπιδοφόρο είναι ότι δεν υπάρχουν ποτέ όρια. Πάντα μπορούμε να ε, φευρίσκουμε διαφορετικές προσεγγίσεις. Κάτι το οποίο με παθιάζει εμένα προσωπικά και οι συνάδελφοι σε εθνικό επίπεδο πάντα αντιδρούσαν ενθουσιοδός ως προς τη δυνατότητα μεγαλύτερης συνεργασίας. Γι' αυτό νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα εμβάθυνσης σχέσεων και θα καταβάλω κάθε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση αν επανεκλεγώ. Ε, Κύριε Μποστινάρη, να απαντήσω άμεσα στην ερώτησή σας. Για τον κοινό μηχανισμό. Θα ήθελα να επαναλάβω ότι εγώ ως ε, διαμεσολαβητής και ο προκατοχός μου έχουμε επωφεληθεί πολύ από την προθυμία της Επιτροπής σας και του Κοινοβουλίου σας να υποστηρίξει τη δράση μας. Και θεωρώ ότι αυτό αποτελεί το σημείο κίνησης. Με άλλα λόγια, η ενίσχυση της περαιτέρω συνεργασίας, προκειμένου να μην κολλάμε στα ίδια, αλλά θα πρέπει να τονίσω ότι η συνθήκη της Λισαβόνας αποτελεί πραγματικά εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη στο σημείο αυτό. Ο διαμεσολαβητής ο Ευρωπαίο διαμεσολαβητής μπορεί να συνεργαστεί σε πολλαπλά επίπεδα με του εθνικού και περιφερειακού ε, συνηγόρου και διαμεσολαβητές. Έχουμε αναπτύξει ήδη ένα σύστημα όπου οι εθνικοί περιφερειακοί διαμεσολαβητές υποβάλλουν ερωτήματα προς τον Ευρωπαίο διαμεσολαβητή για διευκρινήσει, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό δίκαιο και αυτό έχει βελτιωθεί πολύ τα τελευταία χρόνια και τώρα θα ήθελα να ενισχυθεί περαιτέρω αυτή η συνεργασία γιατί η συνθήκη της Λισαβόνας θα ανοίξει και την δυνατότητα διακοινοβουλευτικών επαφών. Δηλαδή, εγώ θα μπορώ να ενθαρρύνω τους εθνικούς ομολόγους μου να έχουν επαφές με τα εθνικά κοινοβούλια και έτσι αυτό το δίκτυο, αν θέλετε, να καταστεί πολύ πιο ζωντανό. Και έτσι, στην πορεία, να τραβήξουμε και την προσοχή των πολιτών πέρα από το θέμα των ετοιμάτων αυτών που υποβάλλονται προς το διαμεσολαβητή, έχουμε χρησιμοποιήσει την ήδη υφιστάμενη δομή του δικτύου. Έχουμε ένα φόρουμ συζήτησης και το οποίο και χρησιμοποιούμε για να δίνουμε συγκεκριμένες απαντήσεις σε συναδέλφους σε εθνικό επίπεδο. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τη δημιουργία του θεσμού του διαμεσολαβητή για θέματα υγείας, σε ό,τι αφορά δηλαδή τους ασθενείς. Κάποιοι ανησυχούν όταν ακούν ότι υπάρχει πιθανότητα να αναπτυχθεί κάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά μέσα από το φόρουμ, μέσα από το δίκτυο ήρθαν και απευθύνθηκαν σε μας, διευκρινίσαμε το θέμα και καταφέραμε να δημιουργήσουμε τέτοιες συνεργασίες, συνέργειες, προκειμένου και να επιληθεί το ζήτημα, αλλά και να βοηθήσουμε τους θεσμικούς, ε, τις θεσμικά όργανα να κατανοήσουν τις ανησυχίες που υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει λοιπόν ανάγκη να υπάρξει απαραίτητα ένας κοινό μηχανισμός. Θα ήθελα μάλλον να ενισχυθούν οι ήδη υφιστάμενοι μηχανισμοί, να χρησιμοποιήσουμε τις ευκαιρίες που μας δίνει η συνθήκη της Λισαβόνας, προκειμένου να υπάρχει μια στρατηγική πολλαπλών επαφών συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής, του Διαμεσολαβητή, των άλλων επιτροπών του Κοινοβουλίου, των εθνικών διαμεσολαβητών, προκειμένου να αναπτυχθούν συνεργασίες που τελικά θα έχουν αποτέλεσμα για τον πολίτη. Κύριε Χάνκης, να σας ευχαριστήσω για την ερώτηση που μου κάνατε. Ξέρω από πού προέρχονται οι ανησυχίες σας. Ξέρω ότι στη χώρα σας έχετε διαμεσολαβητή για τις μειονότητες. Συνεργάστηκα με τον κύριο Κάλτενμπαχ όσο διατέλεσε διαμεσολαβητής για τις μειονότητες και ξέρω ότι δυστυχώς το θέμα των μειονοτήτων αποτέλεσε πολύ σημαντικό θέμα στην όλη ιστορία της περιφέρειάς σας. Το γνωρίζω λοιπόν και ως διαμεσολαβητής, αν επανεκλεχθώ, θα κάνω ό,τι μπορώ για να αντιμετωπίσω το θέμα αυτό. Να σας πω ότι και το γνωρίζω το θέμα και με απασχολεί ιδιαίτερα και θα πρέπει να διευκρινίσω και άλλα δύο στοιχεία. Προφανώς, ως Ευρωπαίος διαμεσολαβητής έχω λάβει εξαιρετικά μικρό αριθμό καταγγελιών σε ό,τι αφορά τις μειονότητες. Οι πιο πολλές καταγγελίες που λαμβάνω έχουν να κάνουν με παραβιάσει των, δικαιώμα, των δικαιωμάτων των Ρωμά στα κράτη-μέλη και ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο είναι ότι όλα αυτά τα θέματα δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητά μου, γιατί εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των συναδέλφων μου σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Αλλά αν κατανοήσουμε, αν ερμηνεύσουμε τις μειονότητες υπό την ευρύτερη έννοια, οι ευάλωτες ομάδες δεν είναι μόνο εθνοτικές μειονότητες. Αν λοιπόν το ερμηνεύσουμε έτσι, προφανώς ο διαμεσολαβητής έχει πεδίο αρμοδιότητας σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τη διακριτική μεταχείριση βασιλικία. Έλαβα μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία σε ό,τι αφορά τα παιδιά με ειδικέ ανάγκες που αποτελεί πολύ σημαντικό θέμα και αν θέλετε βαρύνουσας ηθικής σημασίας υπέβαλα και ειδική έκθεση προς την Επιτροπή σας και προς το Ευρωκοινοβούλιο. Επίσης ξεκίνησα μια έρευνα πρωτοβουλίας και μια δημόσια διαβούλευση για τα ευάλωτα άτομα σε ό,τι αφορά τα άτομα με ειδικέ ανάγκες. Ήταν πολύ ευρύ το πεδίο αυτό. Έχουν γίνει λοιπόν πολλές τέτοιες πρωτοβουλίες. Έχω αναλάβει πολλές τέτοιες πρωτοβουλίες και αυτό καταδεικνύει ότι ο διαμεσολαβητής έχει ήδη αναλάβει δράση σε ό,τι αφορά τις ευάλωτες ομάδες, εντός φυσικά πάντα της αρμοδιότητάς μου. Για να απαντήσω λοιπόν στην ερώτησή σας, είμαι έτοιμος, είμαι πρόθυμος να συνεργαστώ με οποιοδήποτε θεσμικό όργανο, με το Ευρωκοινοβούλιο, με την Επιτροπή, με τους συναδέλφους μου σε, ευρωπαϊκό, σε εθνικό επίπεδο, για να καταργήσω αυτή τη δομή των διπλών μέτρων στην οποία αναφερθήκατε. Πάντα φυσικά εντός των περιορισμών που μου επιβάλλουν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Κύριε Διαμαντούρο, θα ήθελα να, είσαστε, να συγκεφαλαιώσετε περισσότερο και δυστυχώς δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουμε να προωθήσουμε τη διαδικασία ΚΑΣΤΕΑΗ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πάντα είναι το πρόβλημα, αυτό το συνηθισμένο πρόβλημα. Προσπαθούμε να είμαστε συνοπτικοί και να αναφέρουμε τα πάντα, αλλά τελικά δεν έχουμε χρόνο, κυρία Γκούντς. Μιλήσατε για την μείωση του αριθμού των καταγγελιών. Ασφαλώς και μείωση των αριθμών των καταγγελιών και, όπως σας είπα, τρεις μήνες ε, παίρνει η αντιμετώπιση της πιο απλής καταγγελίας. Και να μην ξεχνάτε ότι έχω και 23 γλώσσες πάντα να λάβω υπόψη μου. Προσπαθώ λοιπόν να μειώσω το χρόνο απάντηση στι ε, στις καταγγελίες των πολιτών και ελπίζω να το πετύχω. Κυρία Γουάλης, σας ευχαριστώ και βρίσκομαι υποχρονική πίεση. Το θέμα της κοινή πύλης. Ασφαλώς κυκνηθήκαμε προς την κατεύθυνση αυτή. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα είναι η δημιουργία ενός διαδραστικού οδηγού που δημιουργήθηκε στην αρχή του έτους στα πλαίσια της ιστοσελίδας μας. Μέσω αυτού του οδηγού λοιπόν, ο πολίτης μέσω απαντήσεων και ερωτήσεων θα μπορέσει να κατευθυνθεί προς τη σωστή κατεύθυνση. Άρα ναι, αυτή η κατεύθυνση είναι η κατεύθυνση προς την οποία κινούμαστε. Συμμετέχουμε και στην διαδικασία, αν θέλετε, απάντησης τηλεφωνημάτων. Αν θέλει δηλαδή ο πολίτης μπορεί να λάβει άμεση απάντηση, χωρίς καθυστέρηση. Σε ό,τι αφορά τη Λισαβόνα και το Συμβούλιο και την ε, διαφάνεια, ξέρετε ότι έχω υποβάλει προς το Κοινοβούλιο μια ειδική έκθεση η οποία είχε ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη διαφάνεια στο Συμβούλιο και ανυπομονώ ασφαλώς να συνεργαστώ και με το νέο Συμβούλιο εφόσον επανεκλεχθώ και θα ήθελα να χρησιμοποιήσω και τις νέες δυνατότητες της συνθήκης της Λισαβόνας αλλά το Κοινοβούλιο αυτό θα έχει νέε δυνατότητε να συνεργαστεί με πιο μεγάλη διαφάνεια με το Συμβούλιο επίση. Και θα ήθελα να χρησιμοποιήσω και τη δυνατότητα συνεργασία που δίνει η συνθήκη τη Λισαβόνα για συνεργασία λοιπόν με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Κυρία Άουκεν. Καταλαβαίνω τις ερωτήσεις σας, αλλά δεν είναι εύκολο να τις απαντήσω γρήγορα. Να σας πω ότι το άρθρο 298 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ένωσης θα μπορούσε να αποτελέσει μια βάση για την εφαρμογή του νόμου σε ό,τι αφορά περιπτώσεις καλής διαχείρισης και είμαι φυσικά πρόθυμος να συνεργαστώ με την Επιτροπή σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής σας και του Διαμεσολαβητή για να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για τον πολίτη. Αλλά ασφαλώς αυτό αποτελεί τμήμα, αν θέλετε, μια νομοθετικής δράσης, την οποία θα ήθελα να συνδράμω για το πώς μπορούμε να ε, ε, κάνουμε καλύτερη εποπτεία, παρακολούθηση. Νομίζω μέσω της εντατικοποίησης των δράσεων του διαμεσολαβητή. Και αυτό προσπάθησα να σας ε, περιγράψω. Αν επανεκλεχθώ, σκοπεύω να στραφώ όλο και περισσότερο προς τα θεσμικά όργανα και συγκεκριμένα προς τις υπηρεσίες, προκειμένου αυτή η κουλτούρα της εξυπηρέτησης του πολίτη τελικά όντω να αποβεί προς όφελος του πολίτη. Κύριε Τσίσιστε, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλιά σα. Η καλύτερη απόφαση που έλαβα. Μου φαίνεται ότι μία από τις καλύτερες αποφάσεις μου, για να μην σας πω η κατεξοχή είναι καλύτερη απόφασή μου, ήταν η ειδική έκθεση που υπέβαλα στο Κοινοβούλιο για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Ήταν μια στιγμή κατά την οποία μπόρεσα να ασχοληθώ με μια βασική ανησυχία σε κοινωνικό επίπεδο. Παιδιά, ειδικέ ανάγκες, ειδική εκπαίδευση είναι σημαντικά θέματα στην ε, νομική τάξη του, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι μετανιώνω. Θα σας δώσω την απάντηση ότι θα σας δώσω την εντύπωση ότι προσπαθώ να αποφύγω να απαντήσω. Πάνω από μία απόφαση έχω μετανιώσει. Λυπάμαι που δεν μπόρεσα να παρουσιάσω σαφώς τις θέσεις μου στο Κοινοβούλιο σε θέματα που είχαν να κάνουν με τους, τις αποζημιώσεις των βουλευτών, παρότι καταλήξαμε σε πολύ καλό αποτέλεσμα. Απέτυχα όμως να εξηγήσω σαφώς το θέμα αυτό. Αυτό θα ήθελα να το είχα κάνει διαφορετικά. Πώς να θεσμοποιήσουμε την παρακολούθηση. Νομίζω ότι σας έχω εξηγήσει αρκετά πώς μπορώ. Πώς θέλω να το κάνω αυτό. Θέλω να μπορώ να χρησιμοποιήσω το προσωπικό μου, όχι μόνο εμένα, για να θεσπίσω επαφές ε, με την τοπική και περιφερειακή διοίκηση. Ε, κυρία Πρόεδρε, θα μιλήσω ελληνικά τώρα. Είμαστε υπό ασφιχτική πίεση. Ho già detto che Νομίζω ότι ήδη σας απάντησα για το πώς προτίθεμαι να συνεργαστώ με τους εθνικούς και περιφερειακούς διαμεσολαβητές, ε, άρα επιτρέψτε μου να μην το αναπτύξω. Ε, το θέμα της ε, προαγωγής ενός ε, πνεύματος εξυπηρέτησης ε, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο έχω ήδη αναπτύξει και το οποίο θεωρώ ότι πρέπει να αναπτυχθεί βασικά με την εντατικοποίηση των επαφών του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή με τους θεσμούς. Το ότι οι θεσμοί αυτοί δεν είναι εκλόγιμοι δεν μειώνει την ευκαιρία που μου παρέχεται να μπορέσω συστηματικά να συζητάω με το Κολέγιο των Επιτρόπων, με τους Επιτρόπους, με τους Γενικούς Διευθυντές και επίσης με τους άλλους μεγάλους θεσμούς. Το πώς η ε, πολίτες θα μάθουν περισσότερο για τα δικαιώματά τους. Αυτό νομίζω περνάει οπωσδήποτε μέσα από την αξιοποίηση των ευκαιριών που δημιουργεί η Λισαβόνα και μέσα από τα εθνικά κοινοβούλια. Για μένα τα εθνικά κοινοβούλια είναι κρίσιμος μηχανισμός προσέγγισης. Κύριε Σαλαδράκο, τελευταία ερώτηση. Ε, νομίζω ότι ήδη έχω απαντήσει και απλώς να τονίσω ότι και πάλι ότι για μένα η Λισαβόνα ανοίγει πολύ μεγάλες ευκαιρίες και τις οποίες θα ήθελα να αξιοποιήσω εφόσον μου δοθεί η τιμή μιας νέας εκλογής. Ευχαριστούμε. Μπαίνουμε στη διαδικασία Catch the Eye. Η κυρία Ράπτη έχει το λόγο. Κύριε Διαμαντούρο, θέλω να σας συγχαρώ για τα μέχρι τώρα πεπραγμένα και θέλω να σας συγχαρώ και για κάτι ακόμη. Για την πληρότητα των απαντήσεών σας, αλλά κυρίως για την ειλικρίνεια που διέκρινε τις απαντήσεις σας. Ε, δύο πράγματα μόνο Απαντώντας στην ερώτηση για το τι θα πρέπει να κάνουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα προκειμένου να διασφαλίσουν καλύτερες ε, υπηρεσίες στους Ευρωπαίους πολίτες, επισημαίνεται έξι σημεία, ανάμεσα από τα οποία εγώ ξεχωρίζω δύο. Το πρώτο είναι η ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα δικαιώματά τους και τον τρόπο προάσπισης των δικαιωμάτων αυτών. Και το δεύτερο είναι η παροχή εξηγήσεων για το έργο τους σε γλώσσα κατανοητή για τους πολίτες. Είναι δύο σημεία καθοριστικά κατά την ταπεινή μου γνώμη, γιατί μέσα από τη δική σας δουλειά μπορεί να προαχθεί κατά αποτελεσματικό τρόπο αυτό που συνηθίζουμε να λέμε γενικά, αλλά που έχει ιδιαίτερο ειδικό ενδιαφέρον, η ευρωπαϊκή ιδέα. Και επειδή ε, βλέποντας τα πεπραγμένο σας και ακούγοντας τις τεκμηριωμένες και ειλικρινείς, επαναλαμβάνω, απαντήσεις σας, ε, περιμένω πάρα πολλά από σας και ελπίζω. Να, να δηλώσω ε, και εγώ με τη σειρά μου στους συναδέλφους εδώ της Επιτροπής ότι με την περίπτωση της εισήγησης για την έκθεση του κυρίου Διαμαντρού το 2008 ε, εξάντλησα τα όρια της αντικειμενικότητάς μου. Και χαίρομαι ιδιαίτερα ότι είχα την εξαιρετική τιμή να λειτουργήσω όχι ως Ελληνίδα πέραν της έναν Έλληνα, αλλά ως ένα μέλος ε, ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ανέλαβα την υποχρέωση να εισηγηθώ για ένα άλλο όργανο θεσμικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο εντελώ συμπτωματικά έτυχε να είναι Έλληνας και για το οποίο πραγματικά τώρα μπορώ να σας πω πόσο καμαρώνω που ε, ανέλαβα αυτή την τεράστια ευθύνη. Θα τελειώσω με μία ερώτηση, κυρία Διαμαντούρα. Μιλήσατε κάπου και διαβάσαμε και, στις, ε, και στην έκθεσή σας για τις αυτεπάγγελτες έρευνες. Σε ποιους τομείς θέλετε να μας πείτε πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και την κυρία Ράπτη και την κυρία Παλιαδέλη για τα καλά τους λόγια. Ευτυχώς επειδή δεν έχει πολύ φως δεν φαίνεται πόσο έχω ερυθριάσει με τα υπερβολικές, υπερβολικές Αλλά τις ευχαριστώ παρά τα αυτά. Σε ό,τι αφορά την κυρία Ράπτη, ε, να πω ξεκάθαρα. Θεωρώ ότι είναι απέτηση ενός από έναν όμπουτσμαν να είναι ειλικρινής. Και άρα εκείνο το οποίο κάνω είναι προσπαθώ να ανταποκριθώ στις προσδοκίες του θεσμού, όντας ειλικρινής, αλλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ό,τι αφορά την απλή γλώσσα, θεωρώ ότι και πάλι ο Ombudsman έχει τον, ε, την υποχρέωση να μπορεί να επικοινωνεί με τους πολίτες σε γλώσσα η οποία είναι κατανοητή. Και γι' αυτό έχω επιχειρήσει και έχω απλοποιήσει και τη γλώσσα των αποφάσεών μου και τη ετήσια έκθεση και θεωρώ ότι αυτό πρέπει να επεκταθεί ακόμα περισσότερο και το έχω και εσωτερικά στο θεσμό εφαρμόσει και ευελπιστώ να το εφαρμόσω ακόμα περισσότερο εάν μου δοθεί ευκαιρία να το κάνω. Σα ευχαριστώ για αυτέ τι δύο παρατηρήσει. Σε ό,τι αφορά τέλο την κυρία Παλιαδέλη, κοιτάξτε, οι αυτεπάγγελτε έρευνε είναι ένας πάρα πολύ, ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τον α, διαμεσολαβητή. Πρέπει να χρησιμοποιείται λοιπόν με φιδό και πρέπει να χρησιμοποιείται για κέρυες ευκαιρίες. Οι κέρυες ευκαιρίες μπορεί να είναι είτε αυτό που λέμε συστημική κακοδιοίκηση, δηλαδή πολλά φαινόμενα σε ένα θεσμό το οποίο μας οδηγούν να το κοιτάξουμε, είτε παραβίαση ενός θεμελιώδους δικαιώματος, έστω και από ένα άτομο. Με αυτόν τον τρόπο έχω λειτουργήσει τα τελευταία χρόνια και αυτόν τον τρόπο υποτίθεμαι να λειτουργήσω και στο μέλλον. Δηλαδή να κάνω χρήση τη αυτοπάγγελτη έρευνα προκειμένου να αναδείξω προβλήματα συστημικά και να βοηθήσω να, αν θέλετε, να διαπαιδαγωγήσω του θεσμού πάλι προ την κατεύθυνση τη έννοια του πνεύματο και του πολιτισμού εξυπηρέτηση προ του πολίτε. Ε, Υπάρχει ένα αίτημα ε, Χάρκιν, εκτός χρόνου, έχουμε δύο λεπτά ή δυνατόν σας δίνω το λόγο, ένα λεπτό σε εσά και ένα λεπτό στον κύριο Διαμαντούρο για να απαντήσει. Χάρκιν. Εντάχει. Καταρχήν θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη γιατί δεν ήμουν ε, εξ αρχής της ακρόασης ε, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν σας τιμώ αλλά έπρεπε να βρίσκομαι αλλού. Πρέπει πολλές φορές να είμαστε πανταχού παρόντες. Θίξατε το θέμα των εξόδων των βουλευτών και έχει μεγάλη ε, σημασία γιατί δεν μπορούμε να, το, να αναφερθούμε σε αυτό αλλού. Μιλήσατε για το κατά πόσο πρέπει να είναι κανείς κατανοητός σε μία γλώσσα. Όχι πάντα στη μητρική γλώσσα όλων, αλλά οι πολίτες δεν ξέρουν πώς λειτουργούν τα θεσμικά όργανα πάντα. Τελείωσε το λεπτό μου. Ξέρω ότι διανύσατε μία απόσταση, έχετε περιτέ, περαιτέρω σχέδια έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι οι πολίτες κατανοούν τις απαντήσεις και ότι σε αυτές τις απαντήσεις δεν υποσχόμαστε στους πολίτες περισσότερο από αυτό που μπορούμε να τους δώσουμε. Thank you very much. I appreciate your comments and I'm... Εκτιμώ το σχόλιο σας και είμαι ευγνώμων για το ότι αναγνωρίσετε το θέμα των επιδομάτων των βουλευτών που έθιξα. Ως προς το ερώτημά σας κάθε αυτό, ας σας το θέσω ως εξής. Το εκπληκτικό θέμα της καλοδιαχείρισης είναι ότι είναι ανοιχτό. Κάτι το οποίο μας επιτρέπει να είμαστε ιδιαίτερα ενεργητικοί. Ε, άρα Γνωρίζω πολύ καλά ότι δεν πρέπει να υπερβώ ορισμένα όρια, αλλά πρέπει να είμαι ε, ιδιαίτερα ενεργητικός και να διαδραματίσω ενεργό ρόλο σε αυτό το τομέα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μου είπατε ότι θα πρέπει να εξισορροπήσω, να μην έχουμε υψηλές προσδοκίες και χαμηλές αποδόσεις. Συνήθως συμβαίνει το αντίθετο προσπαθώ να υπόσχομαι λίγα και να παρέχω πολλά εκεί που μπορώ. Και έτσι προσπαθώ να κινηθώ. Αλλά εκτιμώ τα σχόλιά σας και προτίθεμαι να χρησιμοποιήσω απλή γλώσσα. Βεβαίως η ουρανή είναι το όριό μας πάντα, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να χρησιμοποιούμε τη φαντασία μας και να είμαστε ιδιαίτερα δραστήριοι και ενεργητικοί. Ευχαριστούμε κύριε Διαμαντούρο να σας χαιρετήσουμε και να περάσουμε στον τελευταίο υποψήφιο. Ο κύριος Μονέ. Please, Mrs. Mazzoni. Uh, να καλώσουμε τον κύριο ε, Μονέ, να του δώσουμε χρόνο να εγκατασταθεί. For the next 15 minutes. Μπορείτε να μας κάνετε την ε, εισήγησή σας για τα επόμενα 15 λεπτά.